ξανά θα ξεκινήσουμε στις 9 με 1, 3 με 8.30 και 9 με 12 το βράδυ. Η ημερήσια διάταξη είναι